Καλημέρα σας. Θα μιλήσω ουγγρικά σήμερα. Χειρίζω την έναρξη της συνεδρίασης. Στην μέση διάταξη έχουμε μια προφορική ερώτηση σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Επιτρέψτε μου ε, καταρχάς να δώσω το λόγο στον κύριο Μάλκομ Χάρμπορ για πέντε λεπτά. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας θα πρότεινα να καθυστερήσουμε ένα-δύο λεπτά την έναρξη της συνεδρίασης, γιατί πρόκειται για μια ε, προφορική